Να ξεκινήσουμε εκ νέου τη συνεδρίαση. Έχετε ουσιαστικά τα πρακτικά στη διάθεσή σας της χθεσινής συνεδρίασης. Αν κάποιος ε, θέλει σχετικά το λόγο, παρακαλώ. Αν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά και να περάσουμε στο